Συνάδελφοι, παρακαλώ, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Αναθεώρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Απολογισμός και μελλοντικές προκλήσεις. Η συγγήτρια κυρία Μπερές έχει συντάξει και αποστείλει σε όλους τους συναδέλφους το σχέδιο έκθεσης συνοπτικότατο, διξοδικότατο μάλλον. Ε, έφτασε η ώρα να εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης, γι' αυτό σου δίνω το λόγο, Περβάνς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε, η ανταλλαγή αυτή για το σχέδιο έκθεση που νομίζω όλοι έχουν κοιτάξει και στο πνεύμα των όσων έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, σας προτείνω μία προσέγγιση σε τέσσερις φάσεις. Πρώτον, να λάβουμε υπόψη το τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί στην Ευρωζώνη ως προς τις σημαντικές πρόοδους που έχουν επιτελεστεί από το 2010 με την ε, ανάδυση των, ε, του διπτύχου και του εξαπτύχου μέτρων αλλά και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την πραγματικότητα αυτά που μπορούμε να παρατηρήσουμε στην Ευρωζώνη, δηλαδή μια κατάσταση οικονομική πολύ ανησυχητική, εξαιρετικά ανησυχητική, θα έλεγα από τέσσερις διαφορετικές σκοπιές. Πρώτα απ' όλα αυτό που συχνά ακούγεται, η πτώση της ανάπτυξης είναι σαφώς ανεπαρκής. Δεύτερη, η ο αποπληθωρισμός πρώτων θυρών, τουλάχιστον πολύ χαμηλός πληθωρισμός, πολύ χαμηλότερος από αυτό που έχει ορίσει ως στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και που δεν επιτρέπει ακόμα την παρέμβασή της, αλλά πρέπει να διαρωτηθούμε τι θα γίνει με τις χώρες που είναι ιδιαίτερα ε, χρεωμένες, πώς μπορεί να ε, απαλλαγούν από το χρέος και να ξαναρχίσει η ε, διαδικασία δημιουργίας ανάπτυξης. Και έπειτα το τρίτο στοιχείο είναι η ανεργία με μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και ανάλογα με τις ηλικιακέ ομάδες ή τις κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες. Ένα τέταρτο στοιχείο που έχει τονιστεί ιδιαίτερω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ΟΣΑ είναι η η ένταση στις ανισότητες που βρίσκουμε και παρατηρούμε και στην Ευρωζώνη και αλλού. Κάτι που το παρατηρούσαμε και πριν την κρίση ως φαινόμενο, αλλά που κατά κάποιο τρόπο έχει επιταθεί από την κρίση χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων με τη δική μας την παρότρινση ξεκίνησαν μαζί με τον πρόεδρο Γιούνκερ αυτό το τεράστιο πρόγραμμα και εγχείρημα επενδύσεων και το πνεύμα της έκθεσης επικεντρώνεται στο να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει γεφύρωμα ε, και να γεφυρώσουμε την απόσταση μεταξύ του πνευματικού αυτού προγράμματος που δεν είναι ένα ε, φαινόμενο συγκυριακό, τυχαίο είναι μια πολιτική και οικονομική απόφαση που ελήφθη για να αντισταθμίσει τα κενά της ελλείψης της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης που εν τέλει ασχέτως και πέραν της κρίσης έχει, έχουν συμβάλει στην, στο μεγάλο αυτό έλλειμμα. Στο όνομα των μελλοντικών γενεών ε, που πολύ συχνά τις αναφέρουμε και εκφραζόμαστε στο όνομά του χωρίς να τις εκπροσωπούμε αναγκαστικά, μπορεί να πληγούν πολύ περισσότερο από αυτή την έλλειψη επενδύσεων από ότι από κάποιες ε, παραβάσεις και κάποιες ατασταλίες ως προς το δημόσιο χρέος. Το λέω αυτό για τους κανόνες περιχρέους. Τώρα, οι ενδεχόμενες και οι ενδυνάμει βελτιώσεις. Ε, τρία είναι τα βασικά σημεία ε, γύρω από τα οποία διορθώνεται η έκθεσή μου μετά από τη φάση των διαπιστώσεων. Πρώτα απ' όλα συνειδητοποίηση της ε, όλης ανακοίνωσης για την ευελιξία με τρία σημαντικά στοιχεία που πρέπει να σημειωθούν. Το πρώτο είναι ότι αυτή η ανακοίνωση περί ευελιξίας ζητήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Είναι κατά κάποιο τρόπο κάτι που προκαλέσαμε κι εμείς με το έτοιμά μας το επενδυτικό πρόγραμμα να φτάσει σε αίσιο πέρας, αλλά η δεύτερη παρατήρηση ως προς την ανακοίνωση για την ευελιξία είναι ότι προβλέπει πολλές διατάξεις που είναι ίσως ευνοϊκές και τις καλωσορίζουμε για το σκέλος της πρόληψης του δημοσιονομικού ε, συμφώνου, αλλά αν δούμε το διορθωτικό σκέλος, βλέπουμε το περιθώριο ελιγμών, μας δείχνει ότι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε περισσότερα. Και εδώ φτάνω στην τρίτη μου παρατήρηση, δηλαδή καθότι πρόκειται για ένα κείμενο που στην πράξη θέλει να κινητοποιήσει πρώτα απ' όλα το επενδυτικό πρόγραμμα και τα σχετικά κονδύλια, αλλά όχι μόνον, και γι' αυτό θα πρέπει ο συνάδελφο Ούντο Μπούλμαν στα πλαίσια τη δική μα συνεισφορά στην τοποθέτηση του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα Juncker. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ε, συγχρονιστούμε για να μην αρχίσουμε να είμαστε παράφωνοι σαν ορχήστρα που δεν έχει κουρδίσει τα οργανά της. Έπειτα για την ύπαρξη της έκθεσης αυτής είναι η ρήτρα ραντεβού που είχε προβλέψει ο νομοθέτης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό έγινε όταν εγκρίναμε το δίπτυχο και το εξάπτυχο και είχαμε ε, θέση μια διορία ε, επανεξέτασης στις 14 Δεκεμβρίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρόλαβε και εξέδωσε μια ανακοίνωση λίγο πιο γρήγορα, αλλά πρέπει να σας πω ειλικρινώς ως εισηγήτρια ότι ευνηδιάστηκα, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι κατά βάθο είναι λίγο πρόημο να αποτιμηθεί αυτό ο μηχανισμό. Μα εμεί ε, δεν ρωτήσαμε αν είναι πολύ νωρί ή πολύ αρκά. Πρώτα απ' όλα είχαμε θέσει αυτή την ημερομηνία ω ε, ραντεβού. Η Επιτροπή επίση έχει την εμειρεμηνια ω ραντεβου η επιτροπη επιση εχει την υποχρεωση να καταγράψει και να σημειώσει και να λάβει υπόψη, και αυτό το λέμε εμεί ω την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ήταν λίγο γραφειοκρατική η προσέγγιση τη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσει το μονοπόλιο πρωτοβουλία που διαθέτει ως σημείο αφετηρίας και ίσως εδώ έπρεπε να δει και την ποιότητα του διαλόγου που θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ως συνομοθέτες για να ε, ανοίξουμε παράθυρα προς την σωστή θεώρηση του φαινομένου. Εδώ λοιπόν τρία παράθυρα για τη σωστή θεώρηση νομίζω ότι είναι απαραίτητα. Πρώτα απ' όλα είναι σαν να ε, ε, κυνηγάμε το Άγιο Δισκοπότηρο ε, να αναζητούμε το Άγιο Δισκοπότηρο, αλλά θα πρέπει να δούμε τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών και βεβαίως και συνολικά σε άθροισμα τι γίνεται με τη δημοσιονομική φάση των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λίγο σαν το Άγιο Δισκοπότηρο, γιατί το συζητάμε συνέχεια και το αναζητούμε, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε σημείο να το καταφέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα για την συναθρισμένη δημοσιονομική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο ε, ε, συμπεριλαμβάνοντας το χρονοδιάγραμμά μας τα εργαλεία που ήδη υπάρχουν, που προβλέπονται από το δίπτυχο και επιτρέπουν αυτή τη συναθρισμένη θεώρηση της δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών μελών να την έχουμε. Δεν θέλουμε να βλέπουμε μόνο εκ των υστέρων πώς έχει η κατάσταση, αλλά να έχουμε ένα εργαλείο πολιτικο-οικονομικό. Να δώσω ε, ένα παράδειγμα με μια παρομοίωση. Όταν κάθε κάτω μέλο ε, συζητά για τον προπολογισμό, θέτει στόχου. Θέλει να καταπολεμήσει την ανεργία, να προβλέψει επενδύσει, να κοιτάξει τι θα γίνει με την πολεοδομία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, συζητούν για τον προπολογισμό, το ίδιο κάνουν, αλλά με έναν ε, συγκεκριμένο ομοσπονδιακό προπολογισμό. Εμεί στο ευρώ δεν έχουμε καμία, κανένα τέτοιο προπολογισμό. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι να υπάρξει συντονισμό των δημοσιονομικών θέσεων του καθενό κάτω Και εκεί πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε μια συνάθρηση και να είμαστε από πολιτικής άποψης πιο στρατηγικοί στην πιο να έχουμε μια πιο στρατηγική προσέγγιση. Ε, επίσης για το δίπτυχο και το εξάπτυχο η βελτίωση είναι, που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τις μακροοικονομικές ανισότητες. Έχουμε λοιπόν αυτή την ε, μνήα και τη συνεχή αναζήτηση της ε, συμμετρίας, αλλά αυτή δεν εφαρμόζεται. Υπάρχουν σοβαρότατες προκαταλήψεις και πρέπει ε, να δούμε ότι οι συζητήσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται απομονωμένα με το, κράτος, με το κάθε κράτος μέλος για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσει ή να προβλέψει. Μα το πνεύμα, η ίδια η λογική των μακροοικονομικών ανισοτήτων απαιτεί κάτι πολύ πιο ευρύτερο ως προσέγγιση κάτι πολύ ευρύτερο μάλλον ως προσέγγιση. Για την συνολική ισορροπία της ε, Ευρωζώνης ε, δεν φτάνει το 1 συν 1 ίσον 2, αλλά να αναζητήσουμε και το πολλαπλασιαστικό, ε, την πολλαπλασιαστική διάσταση του θέματος, δηλαδή 1 και 1 ίσον 3. Κάπως έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα. Και η τρίτη παράμετρος είναι ότι για τις ενδεχόμενες βελτιώσεις που έχουμε μπροστά μας, χωρίς να υπάρξει όμως αναθεώρηση των συνθηκών απαραίτητο, είναι ότι έχει να κάνει με την αναθεώρηση των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων. Μετά από την αποτίμηση της κατάστασης της Ελλάδα, όπως θα γίνει, και μετά από τα συμπεράσματα που θα διεξαγάγουμε για την δράση της Τρόικας και το κατά πόσον θα ξαναδούμε ένα από τα νομοθετικά σημεία του διπτύχου, του Τούπακ, διότι αυτό ε, καθορίζει τη λειτουργία της Τρόικας. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Και για το 6 συν 2, αυτό το πακέτο, να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο, το χρέος. Ε, συνειδητοποιώ στο εδάφιο, δεν θυμάμαι ποιο νούμερο, Νομίζω ότι είναι η πιο προκλητική παράγραφος αυτής της έκθεσης που ήθελα να συντάξω σε ε, κλίμα συνολική συνένεση. Αλλά νομίζω το θέμα του χρέου πρέπει να το συζητήσουμε με τρόπο εύληπτο. Και θα πρέπει σήμερα να δούμε κατά πόσον είναι ε, χρέο που μπορεί να εξυπηρετηθεί ή να ε, γίνει ανεκτό βάσει των τόσο αυστηρών μα κανόνων. Νομίζω ότι εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει περιθώριο για συζήτηση. Και τρίτο πυλώνα, ο τελευταίο πυλώνα, αυτόν που ανέφερα και το πρωί, παρουσία του πρόεδρου του Eurogroup, είναι η έκθεση των τεσσάρων προέδρων τεσσάρων συν που θα πρέπει να υποβληθεί για, χωρίς να μπω στις λεπτομέρειες, να σας πω απλώς για μένα προτιμότερο θα ήταν, και το λέω εντύμως, θα προτιμούσα την έκθεση των τεσσάρων προέδρων ή την έκθεση Tyson ή το Blueprint Προηγούμενη θητεία βέβαια, αλλά αυτές είναι τρεις ε, πραγματικές ε, βάσεις για τη συζήτηση την οικονομική και την νομισματική. Δεν έχω καμία αμφιβολία σε σύγκριση με το αναλυτικό σημείωμα που μα υπέβαλε ο κύριο Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνω βέβαια ότι εκεί οι συνθήκε ήταν κάπω ιδιαίτερε, αλλά ε, πραγματικά ε, ευθέω και ειλικρινώ στην έκθεσή μα και με το σύνολο των συναδέλφων και τη συνεργασία του, νομίζω ότι θα πρέπει να καθορίσουμε κάποιου δρόμου για να αναζητήσουμε τα κατάλληλα μαθήματα και διδάγματα. Αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008 ε, για τις αποκλήσει στην Ευρωζώνη που δεν μπορούν να παραμείνουν μονίμως και ότι πρέπει να δούμε τον προπολογισμό του κάθε κατους μέλους και την ε, πολλαπλασιαστική διάσταση ε, μεταξύ των κρατών μελών, όλα αυτά που να ληφθούν υπόψη. Ε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εξήλυσα το χρόνο ομιλία μου και νομίζω ότι είναι η στιγμή να ακούσω του σκιώδει εισηγητές και όλου του συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Ο κύριο Τόιρερ, επειδή έχει πτήσει να προλάβει, μα παρακάλεσε να δώσουμε το λόγο πρώτο. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, άρα έχετε κύριε Τόιρερ αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ καταρχάς για, την... Ε, για το γεγονός ότι μου επιτρέπετε να μιλήσω εδώ πιο νωρίς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία κυρία Περές για μια έκθεση η οποία πραγματεύεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση σίγουρα για τις συζητήσεις μας. Είναι στη φύση των θεμάτων οι διαφορετικές πολιτικές ομάδες να αξιολογούμε διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Φυσικά, το σχέδιο έκθεση της ηγητρίας περιλαμβάνει μια σειρά σημείων τα οποία τα μοιράζεται και η ομάδα των φιλελευθέρων, αλλά πιστεύουμε ότι λείπουν κάποια στοιχεία και ότι υπάρχουν και μια σειρά στοιχείων τα οποία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μας. Θα θέλαμε καταρχά να τονίσουμε πιο έντονα στην έκθεση αυτά που ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τελευταία θητεία πετύχαμε θα σας υπενθυμίσω την νομοθεσία για το Six Pack, του ε, Pack. Κάποιοι αμφισβητούσαν το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νομοθέτης θα μπορούσε να είναι σε θέση από τεχνικής άποψης να παράγει μια τόσο σημαντική νομοθεσία. Και εμείς αποδείξαμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Κάποιες προτάσεις ωστόσο που έκανε το Κοινοβούλιο, όπως για παράδειγμα η πρόταση στην έκταση Γκουλάρ για την αυτόματη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη των προδιαγραφών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν ε, εφαρμόστηκαν ε, απόλυτα και αποδυναμώθηκαν ουσιαστικά. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να το υποδείξουμε στο σημείο αυτό, το στοιχείο αυτό. Να αξιολογήσουμε επίσης το κατά πόσον μετά από τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να υπάρχει μια πραγματικά τεκμηριωμένη ανάλυση Πρόκειται για σύντομο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά την επιβολή της νομοθεσίας και σε κάποιες περιπτώσεις καταδεικνύονται θετικές επιδράσεις. Έχουμε την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, όλες χώρες μεταρρυθμίσεων οι οποίες εξελίχθησαν είτε θετικά είτε ουδέτερα και αυτό καταδεικνύει ότι η αποφασιστικότητα για μεταρρυθμίσεις οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα ανάπτυξης από ότι η γρήγορη προσαρμογή της ανταγωνιστικότητας των χωρών σε ό,τι αφορά τις χώρες αυτές. Και υπάρχουν και πολύ σαφή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα η αιτία για την έλλειψη ανάπτυξης είναι η ελλειπής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και όχι οι μεταρρυθμίσεις οι ίδιοι. Επίσης θεωρούμε ότι αν στο μέλλον η Τρόικα δεν θα παίξει με την μορφή αυτή που είχε το ρόλο της, αλλά τα θεσμικά όργανα θα κάνουν τις σχετικές αξιολογήσεις, θα πρέπει να διασφαλιστεί και να εξασφαλιστεί ότι αυτή η ανεξάρτητη αξιολόγηση, αυτή η ανεξάρτητη εκτίμηση των μεμονωμένων χωρών και των αποδόσεών τους θα γίνεται με την κατάλληλη διαφάνεια. Και εδώ πέρα λοιπόν ζητούμε πιο πολύ διαφάνεια, πιο πολύ ανεξαρτησία. Εδώ ο επικεφαλής οικονομικός αναρετής θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Όπως και το αντίστοιχο γραφείο του Κογκρέσου τον ΗΠΑ θα μπορούσε να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τέτοιες αναλύσεις σε ό,τι αφορά τις συστάσεις αναχώρα. Προκειμένου να συζητηθούν όλα αυτά και να συμπεριληφθούν σε μια ανεξάρτητη βάση δεδομένων. Ως ομάδα λοιπόν θα υποβάλουμε μια μεγάλη σειρά τροπολογιών και σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τα στοιχεία που άπτονται της πολιτικής τάξης Πιστεύουμε ότι δεν είναι λειτουργικό το σύστημα, ότι οι αδυναμίες, αν, υπάρχει, αν υπάρχουν, έγκυται στην μη επαρκή και ελαττωματική εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να υπάρχει αξίωση στο μέλλον να είναι πιο συνεπής η εφαρμογή. Το τελευταίο ερώτημα, το θέμα της ενίσχυσης της ανάπτυξης. Εδώ, ναι, οι φιλελεύθεροι θεωρούν ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να ενισχυθεί. Ωστόσο, στο θέμα των εργαλείων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διχάζονται οι απόψει μας και θεωρούμε ότι στο σχέδιο της έκθεσης δεν τονίζεται επαρκώς ότι ω τώρα οι συνθήκε πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιωθούν. Χρειάζεται λοιπόν αποσυμφόρηση από γραφειοκρατικέ προδιαγραφέ και ε, και προβλέψεις για φοροαπαλλαγή για καινούργιες επιχειρήσεις, για κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δοθούν σε κάθε περίπτωση κίνητρα για την ενίσχυση των ιδιωτικών εταιριών, τη διευκόλυνση των ιδιωτικών εταιριών να δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης. Γιατί ξέρουμε ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που απορροφά εργαζόμενους. Τελευταίο θέμα είναι το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρέωσης. Τελευταία φράση για την δημοσιονομική πειθαρχία δεν οδηγεί από μόνη τη στην ανάπτυξη, αλλά ούτε και η χρέωση οδηγεί στην ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να τηρούνται και οι κανόνες για την χρέωση με τους κανόνες που ίσχυαν έως τώρα στο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη με την ευελιξία που προβλέπετε ασφαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λόγια Πρόεδρο. Και τώρα από το ΕΛΚ έχουμε το σκιώδη εισηγητή την Έστερ Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω την εκτίμησή μου για την έκθεση της συναδέλφου Περές. Ξέρω ότι εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ευρύ το πεδίο εφαρμογή τη έκθεση. Και σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι είναι κατεπίγουσα να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Αυτό ισχύει για όλε τι ομάδε. Όλε οι ομάδε αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα τη κατάσταση σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και σε πολλέ περιπτώσεις κοιτάμε την ιστορική διάσταση, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και την εξωτερική διάσταση. Και αυτό ενδεχομένω θα μα λυπεί ακόμα πιο πολύ. Βλέπουμε ότι ο πληθυσμός μας ε, γυράσκει, για... βλέποντας τι γίνεται στην Κίνα με το εργατικό δυναμικό και αναρωτιόμαστε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια ή τι επόμενε δεκαετίε. Και αυτό ίσω είναι πολύ πιο έντονο για τις μελλοντικέ γενιές, τις γενιές των παιδιών μας, τις γενιές των εγγονιών μας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και το ευρύτερο πλαίσιο. Είναι λοιπόν πολύ δικαιολογημένο ότι συζητάμε το θέμα αυτό, αλλά όπω είπατε και συμφωνώ, είναι πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογή τη έκθεση και θα πρέπει να φροντίσουμε η έκθεση να μην ε, επαναλάβει τα όσα είπε η έκθεση για το επενδυτικό πακέτο. Ασφαλώ και χρειάζεται κάποια στοιχεία να τα αναφέρουμε. Αλλά ε, το θέμα του επενδυτικού πακέτου απασχολεί άλλον εισήγητη. Για το ΕΛΚ λοιπόν είναι σημαντικό το εξή. Να σκεφτούμε τις αιτίες ε, που κρύβονται πίσω από τις κρίσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια και τις αιτίες λοιπόν για την προσαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη και για την εισαγωγή του Τούπακ και του ΣΥΚΣΠΑΚ. Συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα βήματα που έχουν γίνει στο παρελθόν τέτοιου είδους συμφωνίες ε, γίνανε σε πολλές περιπτώσεις υπό υψηλή πίεση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως ε, κάποιες φορές να υποτιμήθηκε και να προβλήθηκε πιο πολύ το Συμβούλιο. Ο πυρήνας της ε, έκθεσης ή, εν πάση περιπτώσει, ο πυρήνας του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο και αντιδρούμε, είναι το review clause, η ρήτρα αναθεώρησης. η υποχρέωση δηλαδή στις 14 Δεκάτου του 2014 να εξετάσουμε και να κάνουμε αναθεώρηση του 14 του 6-pack και του 2-pack. Και ποιοι ήταν οι λόγοι που εισήχθη λοιπόν το 6-pack και το 2-pack. Λειτουργήσαν τα νομοθετήματα και κυρίως το βασικό ερώτημα κατά με. Ενίσχυσαν την ε, Ένωση Εποπτείας και την ε, Οικονομική Ένωση σε ό,τι αφορά θέματα χρέους και το καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικά για μένα και σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική σταθερότητα, το scoreboard και το καθεξής. Η εφαρμογή είναι ένα άλλο ευρύ πεδίο το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε σε ό,τι αφορά θέματα ευελιξίας δε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με τα θέματα αυτά. Δεν θα ήταν κακό να αναφέρουμε ότι στο αρχικό σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης περιλαμβανόντουσαν κάποια στοιχεία ευελιξίας ήδη. Και η λογική φαίνεται ότι τώρα πλέον είναι η εξή. Θα πρέπει να μείνουμε... Θα πρέπει να γλιτώσουμε το 3% και να το αφήσουμε. Όχι, στις καλές ε, χρονιές είχαμε χρόνια που, που είχαν Υπήρχαν χώρε, κανονικά στι καλέ χρονιέ θα πρέπει οι χώρε να είναι κάτω το 3%, στο 0% ενδεχομένω. Τι θα πρέπει λοιπόν να συμβεί προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευελιξία, αυτό το στοιχείο ευελιξία στι καλέ χρονιέ, να υπάρχει και αυτό το buffer, αυτή η ενδιάμεση ζώνη, αν θέλετε. για τα, γιατί τα, στις χρονιές των παχαίων αγελάδων έπρεπε να φροντίσουμε και για τις ε, εποχές των ισχυρών αγελάδων, από βιβλικής άποψης. Το θέμα λοιπόν ε, της βιωσιμότητας το, του ρόλου των αρχών. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πιο σημαντικό από το θέμα της ευελιξίας. Πιστεύω λοιπόν ότι αν υπάρχουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις και δεν γίνονται απλά οικονομίες για τις οικονομίες, αν υπάρχει πραγματική ουσιαστική μεταρρύθμιση, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται πιο πολύ χρόνος. Αλλά όπω είπε ο Γερούν Ντέσσελμπλουμ σήμερα το πρωί, το θέμα δεν είναι ή θα κάνουμε το ένα ή θα κάνουμε το άλλο. Δεν είναι διαζευτική η δυνατότητα που έχουμε και τα δύο θα πρέπει να γίνουν. Γιατί αν σε αυτό το χρονικό διάστημα ξεφύγει και πάλι το χρέο, δεν καταφέρνουμε τίποτα. Και το ΕΛΚ αρνείται, αρνείται να επιλέξει αυτή τη λύση. Πόσο μάλλον που η βιωσιμότητα της χρέωσης κάποιων κρατών μελών μας προβληματίζει ιδιαίτερως. Θα κάνουμε κάποιες ε, παρατηρήσεις. Αυτά ως λεπτομέρειες. Αυτό που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Και καταλαβαίνω την επιθυμία της ηγητρίας η οποία εκφράζεται και λέει ποια στοιχεία του ευρωπαϊκού συντονισμού θα πρέπει να υφίστανται. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Όχι όμως σε περίπτωση αυτό που θα οδηγήσει να μην αναλυφθεί καμία ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, γιατί το βλέπω αυτό πάρα πολύ συχνά και έχω βαρεθεί. Όλα λοιπόν τα σπρώχνουμε ως ευθύνη στην κακιά Ευρώπη και σε εθνικό επίπεδο δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αυτό λοιπόν δεν επιτρέπεται. Τελευταίο στοιχείο λοιπόν, το οποίο δικαίω και επισημαίνεται, είναι το θέμα της, ε, του ownership, της ιδιοκτησίας. Πώς θα φροντίσουμε ότι δεν θα κάνουμε μόνο εμεί τη συζήτηση αυτή, αλλά ότι η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί με έντιμο τρόπο και στα εθνικά κοινοβούλια. Το τι σημαίνει να είναι κανεί μέλο τη Οικονομικής και Νομισματικής Ένωση, ότι αυτό δεν έχει μόνο ωφέλη, αλλά και υποχρεώσει ότι το να είναι κανεί μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει να τηρεί και κάποιους κανόνες. Σε αυτά θα περιοριστώ, Πρόεδρε. Αυτά ήταν άλλωστε τα πιο βασικά σημεία τα οποία ήθελα να αναφέρω και προσβλέπω στι μελλοντικέ συζητήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από το ECR ο κύριος Λίκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Μπερές και από δική μας πλευράς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εγκάρδια για την δουλειά σας. Εγώ από δική μας πλευράς θα ήθελα να πω ότι περιλαμβάνονται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στην έκθεσή πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία στην έκθεσή σα, ακόμα και αν ε, θα πρέπει να συμφωνήσω με τον κύριο Τόιρερ ότι σε πολλέ περιπτώσει αποκλίνουν οι απόψει μα και δεν συμφωνούμε με κάποια πολλά μάλλον στοιχεία που αναφέρετε. Θα ήθελα καταρχάς να πω γενικά ότι θα ήθελα να σας προειδοποιήσω να μην ε, ε, τραβηχθεί πάρα πολύ αυτή η έκθεση και συμπεριληφθούν πάρα πολλά στοιχεία. Το θέμα της, ε, πολιτούς έκθεσης είναι ποιες είναι οι προοπτικές και οι προκλήσεις σε ό,τι αφορά τα θέματα των οικονομικών πολιτικών και της οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν θα πρέπει να βάλουμε όπως είπε ο κύριος Τόιρερ. Να συμπεριληφθούν ζητήματα για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με την οικονομική διακυβέρνηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να ξαναξεκινήσουμε να μιλάμε για την κρίση επίση, όπω προτείνει η κυρία Λάγκε εκτός και αν θέλουμε να κοιτάξουμε τις ρίζες της κρίσης που έχουν να κάνουν με την ε, μην τήρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Για τη Lehman Brothers. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία βάση δεδομένων, ε, μία καταγραφή της κατάστασης. Και αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει στην έκθεση. Είναι πολύ επικριτική η έκθεση για την οικονομική διακυβέρνηση, αλλά δεν βλέπω ανάλυση δεν υπάρχει ανάλυση, δεν υπάρχει μια σαφή τοποθέτηση για τα αίτια της μη τήρησης, της μη λειτουργίας των κανόνων του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Και γιατί, γιατί είναι αδιαφανείς και πολύ περίπλοκοι οι κανόνες. Συμφωνώ με την ε, εισηγήτρια ότι το σημερινό οικονομικό πλαίσιο είναι υπερβολικά περίπλοκο και δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτό από πλευρά εθνικών κρατών μελών και των κυβερνήσεών τους. Σύμφωνο επίσης ότι οι συστάσεις οι οποίες γίνονται γίνονται εν μέρη βάσει εσφαλμένων αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό. Γιατί γίνεται αυτό και πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε. διαφωνώ επίσης με την εισηγητρία κάθετα που λέει ότι τα ασφάλματα της ε, σημερινής οικονομικής διακυβέρνησης μπορούν να διορθωθούν με την ε, ε, συνοπτική οικονομική μέθοδο συντονισμού. Πιστεύω ότι αυτό είναι εντελώς λάθος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για συμβατότητα κινήτρων σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων μας και να μιλήσουμε και για μηχανισμούς εφαρμογής και αυτό απουσιάζει παντελώς από την έκθεση. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό το γεγονός ότι η έκθεση δεν εστιάζεται στους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά επεκτείνεται υπερβολικά για το κατά πόσον είναι ευκταίες κάποιες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης κρίσεων στην Ευρωζώμη. Μηχανισμοί δηλαδή και μέτρα αντιμετώπισης ε, κρίσεων για τον αποπληθωρισμό στην Ευρωζώμη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη έκθεση. Εδώ πέρα θα πρέπει να μιλήσουμε για τους κανόνες, τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύσουν μακροπρόθεσμα και όχι να συζητήσουμε συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα για την καταπολέμηση μιας συγκεκριμένης κρίσης. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία απουσιάζουν στην έκθεση. Το ένα έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα των κρατικών χρεών στην Ευρώπη για την εξέλιξη της κρατικής χρέωσης και κατά πόσον αυτή είναι βιώσιμη. Ούτε μία λέξη σχεδόν δεν αφιερώνεται στον τομέα αυτό. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εντελθωθεί αυτό. Και θα πρέπει φυσικά να γίνει αναφορά στο άρθρο 125, το οποίο και αυτό ίσα ίσα που αναφέρεται θα πρέπει να είναι αυτός ο τελευταίος στόχος της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτή η ρήτρα αρρωγής Επίσης, δεν ε, βλέπω τίποτα από τις ε, ακροάσεις των τεχνογρατών, των επιγραγνωμόνων που είχαμε. Ακούσαμε πολύ επικριτικές ε, απόψεις ότι δεν μπορούμε να διακρίνουμε ανισορροπίες σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείμματα ισολογισμών απόδοσης γιατί η εξαγωγή του κεφαλαίου ενδεχομένω να είναι για παράδειγμα ένας ε, σκόπιμος τρόπος για τις επενδύσεις ε, και να εξισορροπηθούν οι εισαγωγές κεφαλαίου. Τίθεται το ερώτημα του κατά πόσον μπορούμε να διαπιστώσουμε από στατιστικής άποψη ε, σωστά, κατά πόσον από οικονομικής άποψης ξέρουμε γιατί μιλάμε όταν μιλάμε για μακροοικονομική ανισότητα. Και κλείνοντας, δεν υπάρχει και αναφορά για το πώς η περιπλοκότητα των κανόνων που υπάρχουν σήμερα και την οποία δικαίως επισημαίνει η συγγύτρια και επισημαίνει και την αδιαφάνεια, πώς λοιπόν αυτή η περιπλοκότητα μπορεί να περιοριστεί. Έχω διαβάσει πάρα πολλά για επιπρόσθετους κανόνες, για επιπρόσθετο συντονισμό, για κοινή ίδια μόρφαση της νομοθεσίας στην Ευρωζώνη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τίποτα δεν βλέπω για την μείωση της περιπλοκότητας. Και λοιπόν, εδώ Πρόεδρε, θα κλείσω όπως μου ζητάτε. Thank Ευχαριστώ. Για την ομάδα του τη Ρίνα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης, την εισηγητρία συγκεκριμένα και για την όλη διαδικασία. Ακούσαμε ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις, ε, όχι απαραίτητα συγκλίνουσες μεταξύ τους και δεν είναι μυστικό να σας πω ότι η ομάδα μας διαφωνεί σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές της ε, διακυβέρνησης. Δεν θα σχολιάσω σημείο προς σημείο το έγγραφο, αλλά θα περιοριστώ στο να επισημάνω τα πιο σημαντικά για εμάς σημεία. Όταν μιλάμε για προσαρμογή στις αιτιολογικές σκέψεις. Εμείς είχαμε πει ευθύς εξ αρχής ότι θέλουμε κοινωνικούς δείκτες. Πρέπει να δούμε τι αντίκτυπο έχει στην ανεργία, στην πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας και το καθεξής. Έχουμε τέτοια στοιχεία και έχουμε γνώσεις που μας δείχνουν πώς άλλαξε αυτή η πολιτική την καθημερινή ζωή των πολιτών και θα θέλαμε να περιληφθούν στις ειδωλικές σκέψεις οι δείκτε εκφράσουμε μια ξεκάθαρη κριτική στην πολιτική γραμμή. Την προηγούμενη εβδομάδα, κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέφερε ότι η τελος παντων αναφερθει οτι υπαρχουν και κοινωνικέ πτυχέ. θεωρουμε επισης οτι θα πρεπει να εκφρασουμε μια ξεκαθαρη κριτικη λιτότητα σε η εξυγίανση έχουν επιπτώσει στη ζωή των πολιτών. Πρέπει να δούμε και πώ επηρεάζει η νέα πολιτική τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι πολλοί, ιδίω στι χώρε σε προγράμματα προσαρμογή, πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει τέτοιε αλλαγέ στην καθημερινή του ζωή που να μιλά κανεί για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική. Δεν μπορούμε να μην Βλέπουμε τι συνέπειες έχει. Από την άλλη πλευρά βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα στα σημεία από 22 έως 25 που λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περισσότερους παράγοντες κατά την αξιολόγηση της κάθε χώρας. Βέβαια, δεν θα πρέπει να βλέπει μόνο τα αποτελέσματα η Κομισιόν. Θα πρέπει να δει και τις επιπτώσεις που έχει για τον άνθρωπο η οικονομική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό για τους απλούς πολίτες Πρέπει ακριβώς αυτό να κάνει η Κομισιόν, να δει τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι πολιτικές στη ζωή των πολιτών. Τώρα, δημοκρατία. Πρέπει να λύσουμε κάποια προβλήματα. Εμείς ε, θέλουμε περισσότερα πράγματα. Θέλουμε και τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν περισσότερο λόγο στις οικονομικές πολιτικές. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι Υπάρχουν αγώνες που πρέπει να δοθούν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των θεσμικών της οργάνων. Θέλουμε σαφείς κανόνες για τα δικαιώματα, τα προνόμια του κάθε θεσμικού οργάνου, για να είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα τόσο για μας όσο και για τους πολίτες. Προσβλέπω και στην υπόλοιπη συζήτηση. Ευχαριστώ. Yeah. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα για την ομάδα FTD, ο Μάρκο Βάλλη. Oh, sorry, sorry. Α, ξέχασα τους πράσινους, ξέχασα. Ο Έρνεστ Ορτασούν Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πρότασή της, κυρίως δε, γιατί δεν ε, υπέκυψε σε πειρασμούς, όπως πολύ συχνά συμβαίνει με τις ε, τοποθετήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν υπέκυψε σε ένα έδος αυτοσυγκατάβασης, αυταρέσκειας και καλής ε, διάθεσης, γιατί ξέρουμε ότι κάτι τέτοια μπάζουν από παντού. Υπάρχει μια κριτική, ένα κριτικό πνεύμα, αυτό διαπνέει την έκθεση και υπό την έννοια αυτή και με αυτό το πνεύμα έχουμε πολλά περιθώρια για να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση και να βρούμε κοινό έδαφος. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι για εμάς είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της νομικής συνόμες αναθεώρησης. Αφήνεται να νοηθεί στην έκθεση ότι υπάρχουν πολλά που δεν λειτουργούν, άρα πρέπει να αναθεωρηθεί το νομικό πλαίσιο στο 2, στο 15, στο 16 σημείο αναφέρονται αυτά. Θα θέλαμε βέβαια ρητό να αναφέρεται το αίτημα για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, διότι αναγνωρίζουμε και εμείς τις ελλείψεις και τις αδυναμίες και δεν θα ήταν λογικό να μην ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μια αναθεώρηση του νομικού πλαισίου. Δεύτερον, συμφωνούμε με την αναφορά που κάνει η συγκήτρια στην ανάγκη περισσότερου εκδημοκρατισμού και περισσότερου ελέγχου εκ μέρου ε, του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Έχουμε και τις συστάσεις αναχώρα. Υπάρχει συναπόφαση μεν για την οικονομική διακυβέρνηση αλλά πολλές φορές ε, τα έγγραφα δεν τα εξετάζουμε τόσο πολύ σε βάθος εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν αναθεώρηση παραλαμβάνω του νομικού πλαισίου για να είναι πιο ε, δημοκρατικό και να υπάρχει δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου ακόμη περισσότερο. θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε ένα θέμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά αυτού του κανόνε, τα πρότυπα, ασκείται κάποια κριτική, όχι βέβαια πάρα πολύ φανή. Ήταν αυτοκαταστροφικά, αυτο, καταστροφικοί αυτοί οι κανόνε, κατά κάποιο τρόπο, οδήγησε ε, η επιβολή του και σε μαζικέ περικοπέ υποτίθεται ότι θα μείωνε αυτό το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης ε, τα επίπεδα του χρέους, ε, τελικά ήταν αυτοκαταστροφικοί οι κανόνες αυτοί γιατί οδήγησαν το αντίθετο σε αύξηση του χρέους και όχι σε μείωσή του. Άρα η οικονομική διακυβέρνηση δεν λειτουργεί. 5. Νομίζω ότι θα πρέπει και το κάνει το κύμα σε έναν βαθμό πρέπει να επιμείνουμε θα πρέπει να αλλάξει η εστίαση πιο πολύ προ τι επενδύσει, δηλαδή, αλλά και στα πρότυπα στου κανόνες διακυβέρνηση να λέμε ότι θα μπορούσαν να τύχουν ειδική μεταχείριση, αν θέλετε κάποιε επενδύσει. Απόσβεση παραδείγματο χαρισμένων επενδύσεων που λαμβάνονται υπόψη στον απολογισμό του ελλείμματο για να υπάρχει μια επιστροφή, μια απόδοση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τα φορολογικά έσοδα. και να καλύπτουν πολλά χρόνια ε, οι διαδικασίες αυτές απόσβεσης. Τώρα, δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε ευελιξία στα πρότυπα και στους κανόνες, μόνο και μόνο όταν έχουμε εκ των πραγμάτων ε, και είμαστε πρώτα τελεσμένου ε, εκτροπές από το πρόγραμμα. Άρα αντικυκλικές πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται πριν την εκτροπή, πριν ε, να έχει γίνει ήδη το λάθος. Να πούμε δηλαδή ότι με χύψη χώρες ε, μπαίνουν σε ύφεση και γι' αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε κάποιους κανόνες ε, μεγαλύτερης ευέλιξης. Πρέπει να αλλάξουν αυτά. Επίσης, η αναθεώρηση της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών το τονίζει το θέμα, το και εμείς. Γιατί χρησιμοποιείται ε, για τις χώρες που είναι σε δυσκολίες, αλλά θα έπρεπε να έχουμε μια πιο γενική θεώρηση και σε ό,τι αφορά τα, τη συμπερίληψη των κοινωνικών δικτών στο scoreboard, αυτό για μας είναι θεμελιώδη σημασία. Και για το δίπτυχο και το εξάπτυχο επιμείναμε και θα επιμείνουμε και ακόμη σε αυτό το σημείο. Επίσης, ε, ολοκληρώνοντας, χρέος το αναφέρει η συγγήτρια και το πλαίσιο διακυβέρνησης ότι πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση, μέρος του χρέους, αυτό είναι σημαντικό. Και τέλος, το ζήτημα της Τρόικας. Ο Γενικό Αγγελέα με την ε, εισήγησή του ουσιαστικά βάζει τελεία και πάυλο στο θέμα αυτό. Κάποιοι προσπαθούν να ε, την αναστήσουν κατά κάποιο τρόπο την Τρόικα, αλλά αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει. Θέλουμε να είμαστε σε ένα κοινοτικοποιημένο ε, πλαίσιο να ε, θεσμοθετημένο. Και η Τρόικα πρέπει να πάψει να υπάρχει γιατί έφερε καταστροφή όπου ε, παρενέβη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Βάρλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Οι σοσιαλιστές ε, και άλλοι συνάδελφοι φαίνεται να θεωρούν ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όμως εγώ ως εκπρόσωπος της ομάδας για την ελευθερία και τη, δημοκρατία, τη συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρώπη πρέπει να πω ότι ως προς την ε, έκθεση αυτή δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο. Ο μηχανισμός της διακυβέρνησης που έχει ε, υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκονται αποτελεσματικό. Βεβαίω, ε, ενδιαφέρον είναι να αμφισβητούμε το δημοσιονομικό σύμφωνο, αλλά αυτό είναι κάτι που έπρεπε να γίνει ευθύ εξ αρχή. Πρόκειται για, κάτι, για κάτι που δεν είναι βιώσιμο. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζουμε έτσι το χρέο. Διότι στραγγαλίζουμε ουσιαστικά, οδηγούμε σε ασφυξία ε, από άποψη δημοσιονομική κάποια κράτη-μέλη. Με το δημοσιονομικό σύμφωνο λοιπόν δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και μετά βλέπουμε τα κράτη να δίνουν μάχη για την ευελιξία που έχει γίνει κάτι και σαν μόδα. Είδατε τι έγινε με τον ε, Τσίπρα που είχε μια κάπως πιο ριζοσπαστική τοποθέτηση. Δεν λέγεται τίποτα για τον υπολογισμό του χάσματος ε, μεταξύ των κρατών. Αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος υπάρχει στο, στην έκθεση μια έλλειψη συνοχής για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Διότι εάν δεν εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση προσεκτικά βλέποντας τι έχει προκαλέσει τις ανισότητες εντός Ευρωζώνης δεν θα καταφέρουμε ουδέποτε να προβλέψουμε ορθούς κανόνες. Θα πρέπει η βούληση του Συμβουλίου να μην περιορίζεται μόνο στην εναρμόνιση της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών. Έχει οδηγηθεί σε κατάσταση μπλοκαρίσματος όλη αυτή η κατάσταση από δεκαετίες, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Και το ευρώ έχει δημιουργήσει σοβαρούς, σοβαρές ανισότητες και στο εμπορικό ισοζύγιο των χωρών, με τη Γερμανία να έχει πλέον να παραβιάζει τους κανόνες με ένα πλεόνασμα που ε, έχει άμεση επίπτωση στην ισορροπία χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και ούτω καθεξής. Ε, εάν λοιπόν δεν αναλύσουμε σωστά την κατάσταση, ε, ενσκύπτοντας τα πραγματικά προβλήματα ανισότητα, δεν θα έχουμε ποτέ ορθούς κανόνες, διότι θα βασιζόμαστε μόνο σε αριθμητικά στοιχεία και παραμέτρους που θα μας οδηγούν κάθε τόσο σε μια οξύτατη κρίση και, της, και κρίση της απασχόλησης και θα αντιμετωπίσουμε διαρκώ τέτοια προβλήματα. Θέλουμε λοιπόν η εξέταση να είναι πολύ πιο ε, επικριτική και μια διεξοδικότερη ανάλυση για το πώς φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση με την οικονομική διακυβέρνηση και τα τελευταία μέτρα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την ποσοτική χαλάρωση και ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας είναι κάτι που θα πρέπει να το συμφωνήσουμε, δηλαδή η ποσοτική χαλάρωση, πώς νοείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με το νόμισμα αυτό και στο σκηνικό της παγκοσμιοποίησης, πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Με συγχωρείτε που ξεπέρασα τον χρόνο μου, ευχαριστώ. Πρόεδρος. Τώρα ε, ο συντάκτης γνωμοδότησης από την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, η κυρία Σιλβί Γκουλάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Περβάνς για την σκληρή δουλειά και όλες τις συνομιλίες που είχαμε τώρα. Κάποιες σύντομε παρατηρήσεις. Έχουμε λίγο δυσκολευτεί εδώ, διότι η οικονομική διακυβέρνηση προβλέπεται στις συνθήκες. Και εφόσον δεν, μάλλον δεν προβλέπεται στις συνθήκες, εφόσον βρισκόμαστε στο δευτερογενές δίκαιο λοιπόν, ε, δεν είμαστε στο επίπεδο που χρειάζεται. Ακόμη και αν έχουμε την πολυτέλεια να προβλέπουμε λεπτομέρειε από την πλευρά λοιπόν τη ΑΦΚΟ, να πω ότι μερικά πράγματα κατά με έχουν να κάνουν και με την αναθεώρηση των συνθήκων. Κατά δεύτερον, και αν θα μπορούσαμε να έχουμε λίγη ησυχία εδώ στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Να πω ότι το σύστημα βασίζεται σε κανόνες, αλλά είναι τελείως ε, γεμάτο ελλείψεις, διότι όταν δεν υπάρχουν απερκείς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, παραλαμβάνει το ΔΕΚ στην Ένωση για, την, ε, ε, για το Δημοσιονομικό Συμφωνό δεν υπάρχει καμία διαδικασία παράβασης ή ακύρωσης για τις αποφάσεις του Συμβουλίου καμία δυνατότητα προσφυγής. Έχουμε ένα σύστημα που δημιουργεί πολύ μεγάλες απογοητεύσεις και όταν λέει ο κύριος Μοσκοβισή ότι οι κυρώσεις αποτυγχάνουν, προφανώς, αλλά οι τι να κάνουν στις χώρες μας όταν εφαρμόζουν τον ποινικό κώδικα. Δεν πρέπει να να αξιοποιήσουν, να κοιτάξουν τις ενδείξεις μιας αποτυχίας και τα αρνητικά περβάνεις, όταν λες για τις μελλοντικέ γενιές είναι πιο σημαντικό να επενδύσουμε παρά να, να προκαλέσουμε και άλλο χρέος. Νομίζω το δημόσιο χρέος, όπως ε, σχεδιάστηκε τα τελευταία χρόνια και σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, γιατί δεν θέλω να μιλήσω για άλλε χώρε, χωρί κανένα σεβασμό τη χρηστή διαχείριση και αυξάνοντα τα τελευταία χρόνια το προσωπικό των αρχών τοπική αυτοδιοίκηση και τα έξοδα, τα τρέχοντα λειτουργία, νομίζω ότι αυτό είναι τελείω ανεύθυνο. Εντάξει, και χρέο και επενδύσει. Σαφώ χρειάζονται επενδύσει, έχει δίκιο, αλλά μιλάμε για επενδύσει που θα χρηματοδοτούνται από καλύτερη διαχείριση των δαπανών. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε στις ε, ωραίες μας, στην ωραία μας χώρα. Ε, επίσης για τις μακροοικονομικές ανισότητες και το λέω υπό τον έλεγχο της ε, Ελίζα Φερέιρα που ήταν η συγκήτρια. Από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούσαμε να αξιοποιήσουμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω ότι είναι ο πιο γόνιμος δρόμος που έχουμε να ακολουθήσουμε. Εάν θέλουμε φιώς να συνδυάσουμε την διαρθωτική προσέγγιση, τη δομική προσέγγιση που να κοιτάζει το σύνολο των προβλημάτων της οικονομίας και όχι μόνο τα χρέη και τα ελλείμματα. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε στην έκθεση ό,τι αφορά αυτή τη διάσταση, συν τους κανόνες ε, ελίματος ε, και, περί, και χρέους, είτε διορθωτικά είτε με την επιβολή κυρώσεων. Και να δούμε και τι μπορεί να κάνει το Διεθνές ε, Δικαστήριο για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Λούκας ως ε, πρόεδρος της ομάδας για την καταπολέμηση της φτώχειας τον προσκαλώ να έρθει να δει τι γίνεται με αυτούς που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Βλέπουμε ότι η επίταση των ανισοτήτων συνεχίζεται, αλλά από αυτά που έρχονται με τις μαρτυρίες τους να μας πούν οι άνθρωποι πιστεύω ότι έχουμε αρκετά στοιχεία για να αναλάβουμε σε αυτό το σώμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Στο πες τη δικασία Κατσιά, άρα μπορώ να δώσω στην εισηγήτρια το λόγο, την κυρία Περμάνος Ελίζα. Α, η Ελίζα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Αλλά αν μου επιτρέπετε να φερω δυο δύο-τρία σημεία. Πρώτο, γιατί συνέβησαν αυτά που συνέβησαν. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κύκλοι, κύκλοι στην οικονομία. Όταν δημιουργείται μια νομισματική ένωση, τα μεμονωμένα κράτη-μέλη καταλείπουν τα εργαλεία τα οποία κανονικά έχουν στη διάθεσή τους για τη διαχείριση αυτών των κύκλων. Από την άλλη πλευρά, δεν δημιουργήθηκαν τέτοια εργαλεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν προέκυψε η κρίση σε μια περιοχή ή στην Ευρώπη συνολικά, την Ευρωζώνη συγκεκριμένα, δεν υπάρχει μηχανισμός εξόδου από την κρίση. Μόνο με εσωτερική απομόχλευση, πολύ επώδυνη πολιτικά και κοινωνικά πολιτική και προσέγγιση. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μέσα σε μια νομισματική ένωση, επειδή είναι διαφορετικές οι οικονομίες και για πολιτικούς λόγους, αλλά στην ίδια αγορά έχουμε την ίδια εμπορική πολιτική, το ίδιο νόμισμα, αυτό δημιουργεί σίγουρα ανισορροπίες και αυξανόμενες μάλιστα ανισορροπίες. Το είπε και η Περβάς σε όλη τη διάρκεια λειτουργία της Νομισματικής Ένωσης. Βλέπουμε αυτές τις ανισορροπίες να αυξάνονται. Σίγουρα μπορούν να γίνουν πολλές προσαρμογές, όπως και αν τις αποκαλέσει κανείς. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να αφερθώ είναι η προσαρμογή που έχει ήδη γίνει. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα νομίζω ότι είναι καιρός να μην προσπαθούμε πλέον να κρύβουμε τα πράγματα. Είναι ανεπαρκής η ανάπτυξη, έχουμε αποπληθωρισμό, τεράστια ποσοστά ανεργίας, αυξημένες ανισορροπίες. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά το γεγονός ότι επιμένει αυτή η κατάσταση ενώ άλλες γραφικές περιοχές ήδη εδώ και καιρό βγήκαν από την κρίση. Η κρίση ξεκίνησε το 8 και βρισκόμαστε στο 15. Οι μεταρρυθμίσεις ίσως δεν πήγαν πολύ καλά και υπάρχουν και άλλα ε, μέτρα τα οποία χρειάστηκε να ληφθούν λόγω της αποτυχίας προσαρμογής. Μετά αναφέρουμε φανταστικά αποτελέσματα σε κάποιες χώρες. Δυστυχώς δεν θα συμφωνήσω διότι ναι υπάρχει βελτίωση σε ένα στοιχείο, δηλαδή στο έλλειμμα και υπάρχει βελτίωση στην πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση. Και αυτό αφού η έκτη είπε ότι θα παρέμβει και θα ελέγξει την κερδοσκοπία πάνω στο κρατικό χρέος, στο δημόσιο χρέο. Υπάρχει όμως τεράστιο χρέος, υπάρχει τεράστια ανεργία, η μεσαία τάξη αφανίστηκε, επενδύσεις μηδέν, και οι ειδικευμένοι οι άνθρωποι με προσόντα αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί σίγουρα μπορεί να έρθει ένα τσουνάμι και μετά αν επιβιώσεις μπορείς να αναπτυχθείς. Το θέμα είναι να επιβιώσεις όμως. Αν έχουμε χάσει το 7% του ΑΕΠ μέσα σε δύο-τρία χρόνια στην Πετσερά στο 26% του ΑΕΠ θέλει πάρα πολύ χρόνο για να έρθει κανείς ε, εκεί που ήταν πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Να είστε λοιπόν πάρα πολύ μετριοπαθείς και συγκρατημένοι όταν αναφέρετε στα δική αυτή ως επιτυχία. Δεν δίνουμε τις σωστές απαντήσεις για τους πολίτες. Δεν είναι απλή απάντηση, είναι πολύπλοκη. Πρέπει όμως να προσέξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και σε ό,τι αφορά τη διάγνωση που κάνουμε και σε ό,τι αφορά λύσεις που προτείνουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ και τώρα. Σα ευχαριστώ και τώρα Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλου του συναδέλφου γιατί πιστεύω ότι ήταν χρήσιμη η όλη συζήτηση. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλέ δυνατότητε να γεφυρώσουμε τι διαφορέ μα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια έκθεση συνεκτική για να μην μείνουμε στην ξύλινη γλώσσα ή να φανούμε αυτάρεσκοι. Δεν μα το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση αυτό. Θα πρέπει να αποστείλουμε σαφή μηνύματα, αν και υπάρχει ένα σημείο στο οποίο νομίζω ότι υπάρχει βαθιά διαφωνία μεταξύ μα και πρέπει να το ονομάσω, να το κατονομάσω. Δεν πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε μεταξύ μας τρόπον την ε, παραπέμπει σε αυτό που είπε ο κύριος Τόλογιαν το πρωί στην ε, ε, ομιλία του απευθυνόμενο στον κύριο Ντάισελμπλουμ. Στους κανόνες μας, δεν λέω ότι ήταν σωστή, έστω στους κανόνες μας, αυτούς που είχαμε, υπήρξε σωστή εφαρμογή ή τα προβλήματα προέκυψαν για άλλους λόγους. Ειλικρινώς δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συνοψίσουμε την οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης σήμερα λέγοντας ότι εφαρμόστηκαν ε, πλημελώς ή κακώς οι κανόνες. Είτε πριν είτε μετά το δίπτυχο και το εξάπτυχο. Δυστυχώς είναι απλουστευτικό να το σκεφτούμε έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να υπερβούμε λίγο τα στοιχεία διαφωνίας μεταξύ μας και από αυτού του κλίματος να εργαστούμε για να είναι επικοδομητική η δουλειά μας. Ως προς την πρόταση Τόιρερ να ενισχύσουμε το λόγο των επικεφαλής οικονομικών της Επιτροπής, εκεί πιστεύω ότι μπορούμε όντως να προχωρήσουμε και να επεξεργαστούμε την ιδέα. Την κρατάω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι πολύ καλή πρόταση, αλλά και πάλι δεν συμμερίζομαι την υπόλοιπη σκέψη, ότι δηλαδή επειδή οι μεταρρυθμίσεις, ότι μάλλον οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν ήταν σωστές, αλλά όχι σωστά εφαρμοσμένες. Δεν αρκεί αυτό για να εξηγήσουμε την κατάσταση. Όσο για τις παρατηρήσεις της κυρία Λάγκε, θα συμφωνήσω και εγώ με την κατεπίγουσα ανάγκη να προχωρήσουμε αυτόν τον τομέα, σωστά την υπογραμμίζει, αλλά φαντάζομαι ότι συμφωνεί μεταξύ μου, μαζί μου μάλλον, ότι σε αυτή την κατεπίγουσα ανάγκη πρέπει να διακρίνουμε και μακροπρόθεσμου στόχου, που δεν είναι λιγότερο επίγοντε το θέμα που καλύπτει η έκθεση των τεσσάρων προέδρων δηλαδή εάν δεν υπάρξει μια σηματοδότηση του δρόμου για εκεί, με προχειρότητες και μαστορέματα θα παραμείνουμε σε διαδικασίες και μηχανισμούς που περιπλέκουν τελικώς την όλη προσπάθεια. Το κοινοβούλιο να καμαρώνει ή όχι για το τι έκανε, αυτό είναι κάτι που δεν θα με βρείτε να διαφωνώ. Ίσως αν θέλετε να προσθέσω και κάτι για να το πω πιο ξεκάθαρα με κάποιο εδάφιο, αλλά δεν είναι το πιο δύσκολο τμήμα της έκθεσης αυτό. Ε, όσο για το θέμα που έθιξε η κυρία Ντελάνγκια για το 3% ή το 0,3%. Για το 0%. Νομίζω εκεί και οι οικονομολόγοι δεν έχουν μία και μόνη απάντηση. Τι θα πει να έχουμε στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο 0% στόχο. Έχουμε μάλλον πάει στην ιδέα του 3% που ταιριάζει πιο πολύ με μια κοινωνία η οποία τουλάχιστον επενδύει λίγο. Για τους στόχους του, για τις συνθήκες του συντονισμού νομίζω ότι εδώ θα έχουμε πραγματικά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ως προς τις παρατηρήσεις του κυρίου Λούκα θεωρεί ότι η έκθεση δεν είναι αρκετά διεξοδική. Να διαβάσω με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις του λοιπόν. Δεν θέλω να τον παραπέμψω στην έκθεση Λίζα και στις λεπτομέρειες που εκείνη περιείχε, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία που χρησιμοποίησα από εκεί για να φωτίσω τη δική μου δουλειά. Και θα διαφωνήσω και σε κάτι μαζί του, εκεί που είπε ότι Αντί να ανησυχούμε για την εφαρμογή των κανόνων, ε, θα έπρεπε να ασχολούμε με τη διαχείριση των κρίσεων. Νομίζω ότι και τα δύο πρέπει να γίνουν. Για την βιωσιμότητα του χρέους έχω εκφραστεί νομίζω σχετικά. Και είναι ένα θέμα που, όπου κανείς, είτε οι χώρες που σέβονται το κριτήριο του χρέους είτε όχι, κανείς δεν έχει δικαίωμα να το παραμελεί, να το παραγνωρίζει. διότι είναι ένα μέρος του παζλ. Υπάρχει πολυπλοκότητα ε, και να διαβάσω με ενδιαφέρον τις τροπολογίες σας γιατί έχουμε κοινό στόχο. Απλώς να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος τρόπος να είμαστε κάπως λιγότερο ε, μπερδεμένοι είναι να έχουμε λιγότερους κανόνες και περισσότερη πολιτική. Εάν σε αυτό συμφωνούσαμε, καλό θα ήταν. Θα μπορέσουμε και να προχωρήσουμε. στο συνάδελφο Ουρτασούν και να ολοκληρώσω εδώ. Νομίζω ότι ένα στοιχείο θα πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο στην έκθεση, ό,τι έχει να κάνει με την σύγκληση και την πρόοδο προς τα εκεί. Μεταξύ των οικονομιών της Ευρωζώνης, ένα στοιχείο που ως τώρα το έχουμε λίγο παραγκονίσει ή αποσιωπήσει. Κατά την άποψή μου, το είπα και το πρωί, δεν νοείται το στοιχείο αυτό να απουσιάζει τόσο εμφανώς από τις διάφορες αναλύσεις και μελέτες του Προέδρου της Επιτροπής, ενώ του είχε ανατεθεί ακριβώ αυτή η εντολή, αυτή η θητεία από την Σύνοδο της Ευρωζώνης. Ε, και αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της σύγκλησης, η φορολογία και το λέω για την Ιρλανδία και άλλα κράτη-μέλη, θα πρέπει να βρεθεί στην καρδιά αυτής της ε, ολοκλήρωσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στη Σιλβή Γκουλάρ από την ΑΦΚΟ είχαμε όντως την ευκαιρία ήδη να συνομιλήσουμε για τα θέματα αυτά, πώς να συμπληρώσουμε τους κανόνες με την δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο για τα θέματα οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, αλλά δυσκολεύομαι να φανταστώ πώς μπορεί η οικονομική πολιτική να τυχήσει σε μεταχείρισεις με, την ποινική, με τον ποινικό δίκαιο, ε, με τον ποινικό κώδικα. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί της ότι η εμβάθυνση της διαδικασίας για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, αυτή η κατεύθυνση πρέπει να εξερευνηθεί περισσότερο, χωρίς να ξεχάσουμε και τις προκλήσεις του χρέους και των ελλημάτων. Ιδού, Πρόεδρε, ποιες ήταν οι μου οι αντιδράσεις στα σχόλια των συναδέλφων. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Για το χρονοδιάγραμμα, μισό λεπτό να σας τα πω. Yes, sorry. Okay. Ε, the deadline... Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών έχει οριστεί η Δευτέρα Μαρτίου. 2 το απόγευμα. Θα εξεταστούν στις 6 το απόγευμα. Σημειώστε. 6 το απόγευμα. 23-24 Μαρτίου εξέταση. Ψηφοφορία στις 14 Απριλίου στην, ε, στην ε, Επιτροπή. Και μετά στην Ολομέλεια. Στις 2 Μαΐου. Τώρα να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Καθίστε παρακαλώ, πάρτε θέσεις. Yes, yes, just a second. Can you take seats so... Καθίστε παρακαλώ να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Φέρετε τις κάρτες σας. In the machine. Okay. Αν έχετε βάλει λοιπόν τις κάρτες στο μηχανάκι, να κάνουμε ένα έλεγχο. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Number of colleagues still to vote. Κάποιοι ακόμα δεν έχουν ψηφίσει.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 52 είναι οι κάρτες. Please, collect, take seat. Here one. Καθίστε συνάδελφοι. Check. Did you vote? Okay, good. Ψηφίσατε. Πολύ ωραία. Ολοκληρώθηκε έτσι η δοκιμαστική ψηφοφορία. Και έτσι μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στην ε, ψηφοφορία μας για την έκθεση Ροζάτη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ξεκινάμε με την συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 19. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Για την τροπολογία υπεριθμών 19. Έναρξη. One Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Μα πρόεδρε, πολλοί συζητούν, πολλοί κάνουν φασαρία. Τι θα γίνει. Take seat and stop. Καθίστε παρακαλώ και σταματήστε τα πηγατάκια. Και επίσης μου περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Υπεράριθμος ένα από το ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική B. Υπέρ. Κατά. Σε τμήματα, συγγνώμη, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίζουμε τον 28. Vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 36. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NV1 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την NV1. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. NV2. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της NV2. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. NV2 δεύτερο τμήμα. Υπεράριθμος 1 από το ΕΛΚ. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. NV3. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την NV3. Έναρξη ψηφοφορίας. Από το ΕΛΚ και από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες είναι ένας υπεραριθμός. Τώρα είμαστε εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική D. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Ή. Ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ή 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. NV4. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την NV4. Έναρξη ψηφοφορίας. Περισσεύει πάλι ένας από το ΕΛΚΑ. Δύο περισσεύουν από το ΕΛΚΑ. Και ένας από τους σοσιαλιστές. Και ακόμα ένας από τους ΕΛΚΑ. Από το ΕΛΚΑ άλλος ένας. Από το ΕΛΚΑ. Εξακολουθεί να είναι υπεράριθμο ένα από το ΕΛΚ. περας ψηφορία. ψηφορίας. Πολύ ωραία. Απορρίπτεται. NV5. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Κατά τη NV5. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής F. Έναρξη. Δύο ψήφοι υπεραριθμές από το ΕΛΚ. Μάλιστα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 82. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας για την 82. Πάλι ένας από το ΕΛΚ. Ακόμη. Εντάξει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΕΝΒΗ. παράγραφος 6. Δεν ψηφίζεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σεμιβάστικη G υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σεμιβάστικη H ήτα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά. Άποχες Α, συγγνώμη, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 101. Πέρας ψηφοφορίας. Μην ασκείτε πιέσεις παρακαλώ στους συναδέλφους. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υποκεφαλίδα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Ι. Άι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ την 118. Ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική J. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται ένβη παράγραφος 9 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Ένδυ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένδυ 11. Υπέρ. Κατά. Είναι κατά εγκουέ. Απορρίπτεται. Ένδυ παράγραφος 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική κάπα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σεμιβαστική L με προφορική τροπολογία υπέρ του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και άρα ψηφίζουμε τώρα το πρώτο τμήμα. Α, όχι. Πολύ ωραία. Συμβαστική μη. M. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 115 υπέρ. 55 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Παραγράφος 13 ΕΝΒΗ. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Έλεγχος, παρακαλώ, για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 13 ένδυ, Έναρξη. Κάποιοι συνάδελφοι ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Μάλιστα. Πέρασε. Απορρίπτεται σεμιβαστική νη. Εν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. σεμιβαστική όμικρον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. σεμιβαστική πι. Ρο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. σεμιβαστική Q. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV14 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. NV15 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Συγγνώμη. Για την NV15 νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέντε συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Δεν θέλουν να ψηφίσουν οι πέντε συνάδελφοι. Καλά. Όπως θέλουν. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. NV16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένδυ 19 πρώτο τμήμα. Παρακαλώ. Σήκωσε τα χέρια. Κατά. 19 πρώτο τμήμα κατά εγκρίνεται. Η γκου ήταν κατά όλοι οι υπόλοιποι. Να, σε, να ελέγξουμε παρακαλώ την ε, NV19 πρώτο κομμάτι, πρώτο τμήμα. Έναρξη. No, they changed part, a group. Άλλαξε, άλλαξε την άποψή ε, μια πολιτική ομάδα. Υπεράριθμο ένα από το ΕΛΚ. ενταξει τη ψηφοφορία ψηφοφορίας τώρα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Έχουμε πρόβλημα συγχρονισμού. Απορρίπτεται. NV20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά έλεγχος για την 180 παρακαλώ έναρξη δύο υπεράριθμοι από το έλκα ένας πέρας Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήταν κατά το έλικα. Α, ήταν υπέρ. Α, ας το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την ε, τροπολογία αρχικού κειμένου. Έναρξη ψηφορίας. Vote is closed. Πέρασε. Close the vote, please. Okay. Yeah. Yes. Adopt. Εγκρίνεται συμβιβαστική R. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 186. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190. Υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος για την 190, έναξη ψηφορίας. Ένας υπεράριθμος, δύο υπεράριθμοί από το ΕΛΚ, πέντε, ψή, ψήφοι λοιπόν. Ωραία, εντάξει τώρα. Ας κλείσουμε την, το, την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Κατά μία ψήφο. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική S. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος για το τρίτο τμήμα έναρξη ψηφοφορία. Δύο υπεράρθμοι από το ΕΛΚ. Ένας. Εντάξει. Πέρασε. Απόρριπτεται. Συμβιβαστική. Ταφ. Υπέρ. Μάλιστα, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη συμβαστική. Την ΤΑΦ, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έγκρινεται. Συμβαστική U. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2.26. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 226. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σεμιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 239 υπέρ κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 239. Ένα ψηφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 240 υπέρ. Κατά. Αυτό ελέγξουμε παρακαλώ για την 240. Έναρξη. Vote is closed. Πέρας. Rejected. 241 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 241. Πέρας. Εγκρίνεται. Ηχή, παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget 2. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την budget 2. Έναρξη ψηφοφορίας. Όπω ξέρετε δεν έχουμε ψήφιση, δεν έχουμε βάλει για ψηφοφορία μια σειρά από τι παραγράφου της Επιτροπή Προεπιλογισμού, γιατί είναι εκτός ε, πεδίου εγκρίνεται. Budget 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάτε τέσσερα πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δεν θα ψηφιστεί. Παράγραφος 5. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ το δεύτερο τμήμα. Νομίζω ότι απορρίπτεται ωστόσο. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6 της Επιτροπής προπολογισμού. Όχι. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Στην παράγραφο 6, δεύτερο τμήμα παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας. Περισσεύει ένα από το ΕΛΚ. Πέρας. Να απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Εγκρίνεται νοούσανε. Ναι. Παράγραφό 8 τη Επιτροπή προπολογισμού υπέρ. Κατά. Άποχες. Η ίδια ισορροπία. Παράγραφος 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος. Έλεγχο ζητείτε. Έναρξη ψηφοφορίας. Παράγραφος 9, έτσι. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Παραγραφός 10, δεύτερο τμήμα παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Παραγράφος 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13, δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 14, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 15 της Επιτροπής Προπολογισμού υπέρ. Κατά. Η φιλελεύθερη είναι υπέρ. Καλά. Εγκρίνεται. Budget 16 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα, αλλά στο ελέγξουμε. Αν θέλετε, για την 16, δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, ας κάνουμε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Πέρας. τα 17 της budget. Υπέρ. Κατά. Η γκου είναι κατά. Απορρίπτεται. Budget 18. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Το δεύτερο τμήμα της 18. Έναρξη. Πέρασε. Απορρίφεται. Συμβιβαστική Y, Y. 19 δεν ψηφίζετε. Γράφει να μην ψηφιστεί και το δεύτερο τμήμα, λέει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 19, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ γιατί δεν βλέπω σαφή διάθεση. Budget 19 δεύτερο τμήμα. Επισήμως, στην επίσημη κατάλογο ψηφοφοριός, αναφέρεται ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική υψηλών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 24, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. σεμιβαστική αλφαβήτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. σεμιβαστική αλφα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18, υπέρ, κατά. Αποχές. Γκουε. Κατά. Έλεγχος. Για την 18. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. λογική σκέψη 1. Στις αναφορές. Να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Αναφορές λοιπόν 1 έως 10. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική Ζ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΑ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Αναφορά 11 έως 15. Unblock. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική κλίση. Έναρξη της ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. 40 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα να περάσουμε στην έκθεση Καϊλή. No, now Ludvigson is after. Now we have first Kylie and then Ludvigson. correct? 30 second breathing time. Okay. <laughs> you change the tires. <laughs> okay. We can start compromise A. Those in Ας ξεκινήσουμε. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά έλεγχος για την 49 άρχεται η ψηφοφορία ε, δύο από το ΕΛΚ είναι υπεράριθμοι Ωραία, πέρας. Εγκρίνεται. Ποια τροπολογία ψηφίσαμε? Τη 49. Και εγκρίθηκε. Τώρα περνάμε στην 50. Να έρχεται η ψηφοφορία. Όχι, με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 50. 50. Vote is closed. Rejected. Compromise B. Τροπολογία Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε για την 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Σι, συμβιβαστική Σι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 72, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε και f υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ κατά Έλεγχος για την 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμμεπαστική G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά Οι σοσιαλιστές δεν βλέπουν να τοποθετούνται. 89 Άρχεται η ψηφοφορία. Στο ΕΛΚ έχουμε έναν υπεράριθμο. Πέρας. Απορρίπτεται. 90. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Έλεγχος για την 91. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε αρχικό κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Στο ΕΛΚ έχουμε έναν υπεράριθμο. Ωραία, πέρας. Απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά Όχι, υπάρχει ένα αίτημα για ξεχωριστή ψηφοφορία για την 108 από τους σοσιαλιστές. Οπότε ψηφίζουμε την 108. 108. Ε, προφανώς ήταν... Ε, υπάρχει αυτό το αίτημα και μπορούμε να ψηφίσουμε ξεχωριστά, οπότε ψηφίζουμε την 108 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 110. Το ίδιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112. Υπέρ. Κατά. Ίδια πλειοψηφία. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική I. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά έλεγχος για την 125 άρχεται η ψηφοφορία έναρξη Πέρας. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική L Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το τρίτο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Ο κύριος Στόλογιαν ανεκτός μικροφώνου. Έχει αποσυρθεί, έχει αποσυρθεί. Η 143. Περνάμε στην 148. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική M, υπέρ, κατά, κατά τμήματα υπέρ, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές 169 169 υπέρ κατά αποχές με συγχωρείτε λάθος λάθος Επαναλαμβάνουμε για την 169. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω αρχικός ε, συνδυασμός ήταν ο ίδιος, αλλά σε ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πάλι στο έλκο είναι περάριθμος ένας. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μία ψηφοδιαφορά. 160... 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. 212 ε, άρχεται η ψηφοφορία. Στο ΕΛΚ έχουμε έναν υπεράριθμο. Πέρας. Με μία ψηφοδιαφορά εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 217. Στο ΕΛΚ έχουμε πάλι έναν υπεράριθμο. Πέρας. Εγκρίνεται. 224. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 218. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμμεβαστική όμικρο. ο, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192. 192 προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Χωρίς την προφορική τροπολογία 192 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται συγγνώμη 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για τη 229. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψηφοδιαφορά. 230 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ. Κατά αποχές Έλεγχος για τη 231. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Ένας. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. 232. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 234. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο αποχές απορρίπτεται, 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 247 υπέρ πρώτο τμήμα μάλλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. W συμβαστική W ε, καταπίπτει 249 από την β. Ε, συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 265 υπέρ μια ομάδα τροπολογιών υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Πάλι ένα υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται μάλλον. Πηγαίνουμε στη συμβαστική X. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 281. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, Συνοδευτική Y υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 287 υπέρ 287. Αποσύρεται. Ωραία. 289. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη 289. Νομίζω ότι γκρίνεται, αλλά στο δούμε. Πάλι ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Ωραία. Πέρας. Με μία ψήφο διαφορά λοιπόν υπάρχει πλειοψηφία. Τώρα περνάμε στην 294 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 295 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 296 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 298 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τιολογική σκέψη α τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Ναι, ναι, είναι άλλη αιτιολογική σκέψη. Έχετε δίκιο. Αρχικό κείμενο αιτιολογική σκέψη τα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρώτη. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ κατά αποχές κρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κα, πρώτο τμήμα ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 31. Έλεγχο. Έλεγχο για τα 30. Ήταν σαφή η πλειοψηφία, αλλά α ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι ένα υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Πέρα. Πάλι ευρεία πλειοψηφία. Κατά. Απορρίπτεται. 31. με συγχωρείτε, 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, πριν να πάω στο 36, διότι εγκρίθηκε η 31. 36 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ συμβαστική 4 κατά τμήματα. Υπέρ, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική, άρχεται ψηφοφορία. Πάλι ένας παράδειγμα από το ΕΛΚ. Και πάλι ένας υπεράριθμος. πέρα ψηφοφορίας, 46 υπέρ, 9 κατά, 5 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση. Ευχαριστούμε. Now we put to the vote. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία του σχέδιου γνωμοδότησης του Μάρκους Φέρμπερ για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, ναι, μπορούμε. Παράγραφος 1, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 1α, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική σ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 46 υπέρ, 11 κατά δύο εποχέ εγκρίνεται η έκθεση και συγχαίρουμε τον κύριο Φέρμπερ, τον εισηγητή. Και περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότηση για την απαλλαγή τη επόμενη υπηρεσία. Παράγραφος 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 1α τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο κειμενο πάραφο 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά ορίστε Πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία. Ωραία, ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαπέντε τώρα, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Καταπίπτει. Έχετε δίκιο και 23. Μάλιστα, άρα πάμε στην τελική ψηφοφορία. Με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 48 υπέρ 11 κατά. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση και περνάμε στην τελευταία απαλλαγή της ΕΣΜΑ. ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τοπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, αρχικό κείμενο. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές,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 Άρα και η γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή κοινωνικών Κινητών Αξιών Αγορών εγκρίνεται. Συγχαίρουμε τον εισηγητή. Ένα λεπτό παρακαλώ μου λένε ότι χρειάζεται. Και μετά να ψηφίσουμε την γνωμοδότηση Λούντβιξον. Άρα διακόπτουμε για ένα λεπτό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Okay, we need updated Α, θέλουμε ένα επικαιροποιημένο κατάλογο ψηφοφορία για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, άρα διακόπτουμε για ένα λεπτό.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 We can start. Everybody's okay. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αν είστε όλοι εντάξει. Συμβαστική Α λοιπόν, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ, κατά, Αποχές. Ήσασταν υπέρ οι σοσιαλδημοκράτες μας. κρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Δ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική I υπέρ I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική K. Περ κατά αποχές Συμβαστική L. Πρώτο τμήμα. Μπορκαρτ. Θέλουμε το έτοιμα για ε, ψηφοφορία κατά τμήματα να το αποσύρουμε. Α, ωραία. Λέω άρα ψηφίζουμε συνολικά την L. VCR όμως. Αποσύρετε εσείς το έτοιμο ή όχι. Επιμένετε. Το αποσύρετε. Όχι. Δεν το αποσύρετε. Άρα ψηφίζουμε. Τέλος πάντων, συνεννοηθήκαμε. Παραμένει ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα τη συμβαστική σέλη. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική M πρώτο τμήμα ονομαστική Ονομαστική για το πρώτο τμήμα. Is roll call voting committee as a, I, as a new? No, there is no rule. No, no, no. There are no rules for roll call votes. But I, of course. Δεν υπάρχει κανόνας λένε για ονομαστικές ισοφορίες, αλλά αν κάποιος ζήτησε να γίνει έλεγχος, είναι μία ή άλλη. Άρα αυτή τη φορά προληπτικός έλεγχος. Για το πρώτο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. κύριος Γκίκολτ. Ίσως να είναι ασύνηθες, αλλά ο κανονισμός δεν προβλέπει ονομασικές ψηφοφορίες στην Επιτροπή. Αλλά δεν με ακούσατε. Αν είχατε ακούσει τι έλεγα, Γκίγκολτ, Σοβαρά το λέω. λένε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ονομαστικές, ενώ μπορούμε. Και λένε ότι είναι έλεγχος. Άρα δεν υπάρχει κανόνας, αλλά δεν απαγορεύεται κιόλα. Ο πρόεδρος, ομολογώ ότι είναι κάτι καινούργιο για μένα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το θέσω ψηφοφορία time if you're just putting it straight in on the day. Yeah, yeah. I like to, I like to sit down and analyze it. I open the vote, so let's open. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε. Αν συμφωνείτε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Πέρας. Μεγάλη πλειοψηφία. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίνεται δηλαδή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Με την προφορική τροπολογία μάλιστα. Α, μάλιστα. Με συγχωρείτε. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα. Προφορική τροπολογία που αποζήτησαν LKCR ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τι θέλετε να ελέγξουμε. Τι έγινε με τον ονομαστική ψηφοφορία.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 αν κατάλαβα καλά, αλλιώ να ελέγξουμε. Τι κάνουμε τώρα, ελέγχουμε την προφορική τροπολογία. Την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία. Πέρασε. Όχι ακόμα. Γιατί ψηφίζουν, ψηφίζουν κι άλλοι. Τώρα μπορούμε. Τώρα μπορούμε να κλείσουμε τη ψηφοφορία. Είστε σίγουρος ότι μπορούμε να περιορίσουμε το μονοπόλιο της, νομοθε... της πρωτοβουλίας από νομικής πλευρά μόνο στην Κομισιόν. Μα ψηφίζουμε ένα κείμενο τώρα, λέει ο Πρόεδρος. Δεν αφορά τη διαδικασία της ψηφοφορίας από το ερώτημά σας. Τι ζητάτε, τι ρωτάτε ακριβώς, δεν κατάλαβα. Κυρία Κουλάρα, απλά λέω ότι εκπλήσωμαι πάρα πολύ που το Κοινοβούλιο βάζει ένα περιορισμό στο μονοπόλιο της πρωτοβουλίας Κομισιόν για τις νομοθετικές προτάσεις. Δεν ξέρω, το δικαστήριο το θεωρεί νόμιμο αυτό. Αλλά ας ψηφίσουν παρόλα αυτά. Πολύ αργά για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις, τα recitals, στο 2. Ψήφι πέρ. Τις τροπολογίες 64 στην αιτιολογική σκέψη 2. Ψήφι υπέρ. 64. Κατά. Αποχές. 64 τροπολογία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 65 καταπίπτει, τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την τροπολογία 66, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Νη. Ψήφι περ. Κατά. Το έλκ υπέρ της 1. Μάλιστα. Εγκρίνεται. Όχι, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι φιλελεύθεροι δεν βλέπω τι κάνουν. Είστε υπέρ κατά. Μάλιστα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Α. Να ελέγξουμε την 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική π. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T ταφ υπέρ υπέρ λέω κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική Γιού, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Ορίστε. Calculated the new number of it's four, not seven. It's four members. The, because uh, it's four. Is the, In roll call vote, the vote is open. Λοιπόν, ονομαστικά ψηφίζουμε, άρχεται ψηφοφορία. The vote is... ψηφοφορίας. 38 υπέρ 16 κατά 5 αποχές. Εγκρίνεται έκθεση συγχαρητήρια στον εισηγητή. So we can conclude... Μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Η ψηφοφορία των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγορά θα γίνει την Πέμπτη το πρωί σε 9. Είναι σημαντική ψηφοφορία να είστε παρόντες. Καλό απόγευμα.